Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Η συγητής είναι ο κύριος Χόκμαρκ. Είναι παρόντες οι σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων. Μπορούμε να αρχίσουμε. Έχετε το λόγο κύριε Χόκμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Η γενική μου κρίση για τις τροπολογίες είναι ότι από πολιτική άποψη τουλάχιστον θα είναι εύκολο να τις ομοδοποιήσω σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Μετά την δημόσια κρόση της 27ης Ιουνίου θα φροντίσω να συζητήσουμε συμβιβαστικές προτάσεις των διαφόρων παραγράφων μεταξύ των σκευδών εισηγητών ώστε να ετοιμαστούμε για την ψηφοφορία στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, η γενική δομή των τροπολογιών, όπως σας είπα, δείχνει μια αυξημένη ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας, γενικής συζήτησης και παγκόσμιου πλαισίου για το τι εννοούμε με την παγκόσμια διακυβέρνηση. Έχουμε τους G20. Πολύ σημαντικό φόρουμ γιατί εκεί συμμετέχουν 20 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου αυτό προσδιορίζεται κατά κάποιο τρόπο το G20, αλλά έχουμε και άλλες παγκόσμιες δομές, τις αναδυόμενες οικονομίες, ε, τις χώρες BRIC και τις πιο παλέμαχες G7 και G8. Πάντως ε, η G20 με τις άτυπες δομές είναι πιο σημαντική. Και ήταν και το βασικότερο φόρουμ συζήτησης για την παγκόσμια διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Αντιμετώπιση της κρίσης, συζήτηση νέων κανόνων και διατάξεων στα πλαίσια της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αλλά διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες στη G20. Η βασικότερη είναι η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη λογοδοσίας, η έλλειψη οικουμενικότητας και πάλι η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη εφαρμογής. Γι' αυτό και στην έκθεσή μου λέω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την G20 με άλλες περιφερειακές δομές και με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο που παρέχει τα εχέγγυα διαφάνειας επειδή έχετε βελτιώσει με διαφάνεια αλλά λογοδοσίας. Οπότε υπάρχουν περισσότερες εγγυησει για αξιόπιστη εφαρμογή. Και όταν διαβάζω τις ε, τροπολογίες διαπιστώνω ότι οι περισσότερες σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων αναφέρονται στις δομές αυτές και στο ειδικό τους βάρος. Οπότε γι' αυτό είπα ότι από πολιτική άποψη θα είναι εύκολο να βρούμε συμβαστικές λύσεις, συμβαστικές τροπολογίες ακολουθώντας αυτή τη δομή. Βέβαια θα προσπαθήσω αν όχι να ικανοποιήσω όλους, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό να βρουν όλοι κάποια ικανοποίηση. Οι τροπολογίες Κλούνα, Τρομόσα, Γκέραρτ είναι εύκολο να γίνουν δεκτές ή να συμπεριληφθούν σε συμβαστικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες Λάμπερτ Διαφέρουμε σε ορισμένα σημεία. Θα το συζητήσουμε. Δεν μας εκπλήσει αυτή η διάσταση απόψεων. Έτσι έχει ζωή. Αλλά τις τροπολογίες 22 και 57 μπορώ να τις δεχτώ. Τις 22 και 57 τις δέχομαι τις δικές σας. Για τις υπόλοιπες θα το συζητήσουμε. Η κυρία Μπερές κατέθεσε πολλές τροπολογίες. Μερικές πολύ ευχαρίστως να τις δεκτώ αυτούσιες. Πάντως είμαι συνεργάσιμος, θέλω να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Για τις παραγράφους, το σημείο 4 είναι σημαντικό. Αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Και τα νομίσματα που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το, στα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κυρίως ε, αναφερόμαστε εδώ στο κινέζικο πρόβλημα. Γιατί αν θέλουν ορισμένες χώρες ε, να μπουν τα νομίσματά τους στα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα του Δουνουτού, θα πρέπει να είναι μετατρέψιμα αυτά τα νομίσματα. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Μετατρέψιμα μετατρέψιμο κινέζικο νόμισμα. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Τώρα, οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου. Ας το αφήσουμε αυτό κατά μέρο. Έχουμε κάποιες άτυπες δομές και του G20, αλλά και άλλων περιφερειακών οργάνων. Το αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε αξιοπιστία, σταθερότητα, να εξασφαλίσουμε εφαρμογή σε συνδυασμό κατά κάποιο τρόπο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς θα γίνει αυτή η συνάρθρωση θα το συζητήσουμε με τους ε, σκιώδεις συγκητές. Κυρία Μπέρες, την ώρα που μπαίνατε έλεγα ότι τουλάχιστον ε, δύο τροπολογίες σας πολύ ευχαρίστω θα τις δεχτώ. <laughs> Και χαίρομαι που το λέω γιατί δεν ε, ισχύει πάντα τέτοια αποδοχή. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Χακμάρκ. Γιατί το σχέδιο έκθεσης αποτέλεσε μια πάρα πολύ καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να οικοδομήσουμε και νομίζω τα βασικά υπάρχουν. Και ε, το έχουμε κάνει αυτό και ελπίζουμε τώρα, να αναμένουμε την συζήτηση των συμβαστικών προτάσεων για να γίνει αυτή η έκθεση σημαντική και ισχυρή ε, εισαγωγικά. Πρέπει να πούμε πως η παγκοσμιοποίηση έκανε μεγάλα άλματα την τελευταία δεκαετία και οδήγησε τις ε, αναδυόμενες χώρες στο να αναδυθούν και άρα άλλαξε το τοπίο. Του του δεν μπορούμε να γνωρίσουμε βεβαίω. το τεράστιο θέμα, το ότι υπήρχε οικονομική κατάρρευση που ακολουθήθηκε μετά από μία μεγάλη ύφεση από την οποία ακόμα υποφέρουμε, δεν έχουμε δει ακόμα το φως στο τέλος του τούνελ και επίσης παρά το ότι είδαμε κάποιες ε, ανερχόμενες χώρες να εμφανίζονται, κάποιες έγιναν ακόμη φτωχότερες. Και υπάρχουν βέβαια και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ουσιαστικά νομίζω πως, όπως είπε ο κ. Χόκμαρκ, έχουμε τα θεσμικά ζητήματα και μετά τα υπόλοιπα ζητήματα, δηλαδή σε θεσμικό πλαίσιο και σε πλαίσιο παγκόσμιας λήψης αποφάσεων ε, πρέπει να δούμε τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι είδου διακυβέρνηση θέλουμε. Έχουμε τους G20. Θέλουμε να αλλάξει και να γίνει άλλος ένας ΟΗΕ όπου θα συζητιούνται πράγματα και δεν θα συμφωνούμε ποτέ ή θέμε μια λέσχη όπως είναι τώρα, μεγαλύτερη μεν όπου οι ισχυρότερες χώρες εκπροσωπούνται και οι BRIC οι λεγόμενες αλλά οι μικρότερες και φτωχότερες δεν έχουν φωνή. Τι θέλουμε λοιπόν ακριβώς. Μια επιτυχία είναι αυτή. Μετά. Πόσο οργανωμένοι πρέπει να είμαστε. Το γεγονός ότι λαμβάνουμε αποφάσεις με συνένεση σημαίνει πως καταλήγουμε με ανακοινώσει τύπου τόσο αφηρημένε που δεν σημαίνουν τίποτα. Και δεν υπάρχει μετά καμία συνέχεια έτσι ώστε να ξέρουμε εάν ε, έγιναν τα όσα υποσχόμαστε. Ποιο ήταν ο ρόλο επίση των G20 σε σχέση με διεθνεί οργανισμού, ε, Δονοτού, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΣΑ. Θα θέλαμε να δούμε κάποια σχέση μεταξύ αυτών και των G20. Και στους G20 βεβαίως ε, έχουμε μια ισχυρή γραμματεία που δεν υπάρχει. Αν πάτε στο site θα δείτε πως υπάρχουν πολύ ισχυρότερε υποδομέ για άλλους διεθνεί οργανισμούς και λίγες για το G20, πλην των ανακοινώσεων τύπου που βγαίνουν. Μετά, η άλλη θεσμική πτυχή είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μία φωνή που λέμε ότι θέλουμε να έχουμε, που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, με βάση το τωρινό οικονομικό τοπίο. Έχουμε διάφορες φωνές Αλλά δεν είναι αυτό το, το θέμα. Εντάξει, είμαστε ισχυροί, με σεβασμό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, πρέπει να έχει μία φωνή που να ακούγεται ισχυρή. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι αυτό το οποίο έχουμε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ανισορροπίες. Οι είναι οι ίδιες και προκαλούνται από πλεονάσματα από τη μία και ε, λίγη κατανάλωση και το αντίστροφο στις χώρες τις ελληματικές. Ναι, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση και ε, καθόλου επενδύσεις. Θέλουμε λοιπόν συμμετρία, γι' αυτό τονίζουμε και στο επίπεδο της Ένωσης και στο παγκόσμιο επίπεδο το θέμα αυτή της συμμετρία. Το θέμα αυτής της ισορροπίας, ότι για να ανυψωθεί ο ένας πρέπει να μειωθεί ο άλλος, και το ίδιο ισχύει και για την κίνηση βεβαίως χώρες αυτές. Το ίδιο και για την Κίνα και τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άλλα ζητήματα ισοτιμίες συναλλαγματικές ε, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια χωρίς πιέσεις ε, που να ενισχύουν αυτές τις ανισορροπίες. Θέλουμε ένα νέο διεθνές ε, νομισματικό σύστημα, πιο αποτελεσματικό από το τωρινό. Θέλουμε επιτέλους να δούμε ποιος είναι ο ρόλος το που θα πρέπει να έχουν τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Θα πρέπει να συνεχίσει το δολάριο ως έχει, να χρησιμοποιείται ως αποθεματικό νόμισμα ως διεθνές νόμισμα με όλα αυτά τα, τα προβλήματα. που αντιμετωπίζει στη, στη ΣΥΠΑ. Και επίσης θέλουμε συνεπή ρύθμιση χρηματοοικονομική και στις δύο όχθες του Ατλαντικού και όσον αφορά α, προδιαγραφές και λογιστικά πρότυπα και να μην υπάρχει αρμπιτράζ και να διαλέγει κανείς το συμφερότερο ρυθμιστικό καθεστώς. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα. Θεωρώ πως ε, τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν οπωσδήποτε στον κόσμο αξίζει πολύ καλύτερο θεσμικό πλαίσιο και λήψη αποφάσεων και αναμένω τη συζήτηση αυτή τη συζήτηση με τους ε, σκιώδεις συζητητέ ε, και τον κύριο Χέκμαρκ που ε, και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά εργάζομαι, στα αγγλικά επικοινωνώ με τον εισηγητή και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ τον κύριο Χάκμαρκ. Απουσίαζε στην παρουσίασή του σχέδιο έκθεση, αλλά ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την υποβολή αυτή τη έκθεση. Είναι αρκετά ισορροπημένη και εμπεριστατωμένη. Όταν θα προσδιορίσουμε τελική τη μορφή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα αποτελέσματα της Επιτροπής Κρίσης, ώστε να είμαστε συνεπείς στις διάφορες επιτροπές και στα πόρισματά τους. Δεν θα εξετάσω διεξοδικά όλα τα σημεία, θα εμείνω σε ορισμένα θέματα που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Συμφωνώ απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει έδρα σε όσο το δυνατό περισσότερες διεθνείς οργανώσεις. Είμαι υπέρ της ενιαίας έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωζώνη, γιατί χρειαζόμαστε μία ενιαία φωνή αν θέλουμε να έχουμε κάποιο βάρος σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και πολυπολικό. Σε ό,τι αφορά τις τιμίες χρειαζόμαστε ένα νέο νομισματικό σύστημα και να, χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Επίσης θα πρέπει ε, να καταγγείλουμε το νομισματικό dumping που κάνουν ορισμένες χώρες όπως η Κίνα στις αγορές. Γιατί αν δεν το καταγγείλουμε, ίσως δημιουργηθούν αντίστοιχα κίνητρα και σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες να προσφύγουν σε αυτό το dumping του νομισματό τους. Ε, ένα διοικητικό συμβούλιο κεντρικών τραπεζών ίσως ήταν χρήσιμο για συντονισμό νομισματικών πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό και συμφωνώ με την αντίστοιχη τροπολογία του κυρίου Νταφ. σε ό,τι αφορά το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα ήταν χρήσιμο μέσο για την αύξηση των εσόδων στα πλαίσια της αύξησης ε, των επιπέδων δημοσίων χρεών. Συμφωνώ με το φόρο αυτό το χρηματοπιστωτικό συναλλαγών, αρκεί να ισχύσει παντού. Και συμμερίζομαι τις ανησυχίες που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή από τον Μάριο Ντράγκη ε, που εξέφρασε ανησυχίες για την ρευστότητα και την κερδοσκοπία που θα μπορούσε να προκαλέσει η θέσπιση αυτού του νέου νόμου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όπως είπα όμως και στο παρελθόν, δεν θα στηρίξουμε ένα τέτοιο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αν θεσπιστεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θεσπιστεί θα πρέπει να θεσπιστεί παγκοσμίω. Αλλιώ μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα οδηγήσει σε διαρροή κεφαλαίου από την Ευρώπη και δεν θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτή είναι η θέση μου. Ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε και στα πλαίσια αυτής της έκθεσης, γιατί και άλλες εκθέσεις περιστρέφονται γύρω αυτό το θέμα. Τέλος, θα ήθελα να υποστηρίξω και δημοσίως την προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού συντονισμένου πλαισίου χρηματοπιστωτικού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, γιατί όταν λέει πως δεν συμφωνούμε, εγώ αισθάνομαι καλά. Εντάξει, αν συγκλίνουμε σε κάποια πράγματα, ε, εντάξει, εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές διαφορές και βεβαίω αυτό το οποίο θα έλεγα και σε σχέση με εσά και τους φιλελεύθερου αυτό το οποίο δεν πιστεύουμε είναι πως το εμπόριο αυτού θα κάνει αηφόρο την παγκόσμια οικονομία και τη ζωή στον πλανήτη. Οπότε δεν είμαι υπέρ των εμποδίων για τα εμπόδια, δεν είναι καλό αυτό, αλλά από την άλλη δεν θεωρώ πως το εμπόριο χωρίς αυστηρούς κανόνες ε, είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε εμπόριο, χρειαζόμαστε και κανόνες. Γιατί οι αγορές δεν λαμβάνουν αυτά τα οποία λένε εξωτερικότητες οι οικονομολόγοι υπόψη. Πράγματα τα οποία δηλαδή καταστρέφουν τις συνθήκες ζωής είτε κοινωνικές είτε περιβαλλοντικές. Οπότε διαφωνούμε, αλλά βεβαίως ε, περιμένω τυχόν συμβιβαστικές πρωτοβουλίες, έχω εμπειρία συνεργασίας μαζί σας σε άλλα ζητήματα και έχω δει πως κάποιες φορές μπορούμε να συγκλίνουμε. Κάποια πράγματα που θα ήθελα να τονίσω. Συμφωνώ με αυτό το οποίο υπόθηκε για την ενιαία ευρωπαϊκή φωνή στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάτι γενικό για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Το χρειαζόμαστε, το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε πως απέχει πολύ. Και αυτό το οποίο με ανισχύει είναι, όπως είπε ο Ραμόν για τον φόρο αυτόν, τόσο μην αναφερθώ μόνο στο φόρο, όταν λέμε πως θέμε ίσους όρους ανταγωνισμού και πριν σιγουρευτούμε για κάτι τέτοιο δεν θα κουνηθούμε, δεν αναφέρομαι πάλι στο φόρο συγκεκριμένο όπως είπα. Η ιστορία της Ευρώπης και πριν από αυτό η ιστορία της παγκόσμιας οικονομικής τάξης που διαμορφώθηκε από τις συμφωνίες Bretton Woods δείχνει πως μια φορά όταν ε, δεν περιμένει κανείς παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση ξεκινάει με έναν συνδυασμό, με, έναν, με μια συμμαχία των προθήμων γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμμαχία των προθήμων που μοιράζεται την κυριαρχία σε κάποιους τομείς για να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε πως είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Και, και θα έλεγα πως αφενός πράγματι είναι κάτι το επιθυμητό η παγκόσμια και η οικονομική διακυβέρνηση, αλλά δεν θα πρέπει να πιστεύουμε πως θα γίνει σύντομα. Βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι η Ντόχα στους γύρους του ΠΟΕ. Η G20 είναι, συγγνώμη, αλλά είναι ένα πουκάμισο αδιανό. Καλό είναι που υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις, αλλά όσον αφορά πραγματική πολιτική συνένεση έχει αποτύχει. Οι ΙΠΑ έχουν ε, ποσοτική χαλάρωση, οι Κινέζοι ξοδεύουν, οι Ευρωπαίοι λιτότητα, διαφορετικές συνταγές και το μόνο που κάνει το G20 είναι να μιλάμε ο ένας με τον άλλον, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και πάμε σπίτια μας. Μην γελιόμαστε λοιπόν. Ε, η G20 δεν είναι υποκατάστατο για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Χρειάζεται καιρό ακόμα και δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για το να κάνουμε πράγματα εντό των τεσσάρων ε, τείχων, θα έλεγα, τη ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν περιμένουμε και ε, προχωράμε εμείς μπροστά. Λίγα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω τώρα η κινητικότητα των τιμών των βασικών αγαθών. Τώρα ε, βλέπετε είχαμε κάποια ξηρασία στην Ευρώπη, άλλες φορές μπορεί να είναι αλλού. Ξέρετε πως ειδικά τα τρόφιμα και οι τιμές των τροφίμων είναι πραγματικό ζήτημα. Λιγότερο σε, στις χώρες μας παρά περισσότερο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αν θέλουμε λοιπόν παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση να έχει κάποια νομιμοποίηση για τους φτωχότερους αυτού του πλανήτη, Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί τότε θα τους δείξουμε πως ε, είναι και προς το δικό του συμφέρον. Όχι μόνο προς το συμφέρον του ανεπτυγμένου κόσμου. Πράγματι, πρέπει να γίνει κάτι από πλευράς ε, κεφαλαιακών ροών. Δεν λέω πως θα πρέπει να ξαναπάμε στις εθνικές αγορές κεφαλαίου. Αυτό το οποίο λέω είναι πως Έχουμε δει τι έχει κάνει το επίπεδο αλληλεσύνδεσης παγκοσμίων οικονομικών ροών όσον αφορά το πόσο ευάλωτο είναι ολόκληρο το σύστημα και αυτό είναι σοβαρή υπόθεση. Uh, uh, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε στα αγγλικά, αλλά τα διαμερίσματα του πλοίου πλέον δεν διαχωρίζονται από μπουλμέδες είναι μία η δεξαμενή και θα βουλιάξει το πλοίο. Και το πλοίο είναι η παγκόσμια οικονομία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερα στεγανά, διαμερίσματα, για να μην βουλιάξει όλο το πλοίο. Οπότε, αυτό το οποίο με συνάρπασε εμένα ήταν η σημερινή επίσκεψη από την Πρωθυπουργό των Βερμούδων. Ε, ε δηλαδή ήταν αστείο αυτό. Εγώ δεν είχα όρεξη για αστεία σήμερα το πρωί, αλλά το να μου λέει κανείς πως έρχονται στις ε, γιατί έχουμε παγκόσμιο οικονομικό κέντρο, ε, ε, ε, Κάποια άλλη λόγοι υπάρχουν. Και απευθύνομαι εδώ πέρα στους φιλελεύθερους. Δηλαδή, αν μιλάτε σοβαρά για τη μείωση της φορολογικής πίεσης, δεν θα διαφωνήσετε μαζί μας πως το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη. Γιατί αν φόροι, φόροι ε, που οφείλονται καταβάλλονται, δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε νέους φόρους. 300 δισεκατομμύρια υπολογίζεται η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη και αυτό γίνεται μέσω αυτών των φορολογικών παραδείσων εντός και εκτός της Ένωσης. Οπότε αν μπορούμε να πιάσουμε κομμάτι, εντάξει δεν είμαι και βλάκας, μηδενική φοροδιαφυγή δεν θα γίνουμε ποτέ. Γιατί εντάξει, αυτό μετά περνάμε σε αντιδημοκρατικά μέσα και βλάπτουμε τις ε, αστικές ελευθερίες. Αλλά αν μειώσουμε ουσιαστικά την ε, φοροδιαφυγή, νομίζω πως οι προπολογισμοί θα γίνουν ε, πιο υγιείς. Και εκεί πέρα λοιπόν έχουμε πολλά να επιτύχουμε στο πλαίσιο της παγκόσμια οικονομικής διακυβέρνησης. Uh, Συμφωνώ με πολλές τροπολογίες, αναμένω λοιπόν τη συζήτηση. Ελπίζω να καταλήξουμε συμφωνία ή να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε ως συνήθως. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ Φιλίππη, κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας ε, και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα σε όλη, κατα, όλη την ανάλυση των τροπολογιών, αλλά δεν πιστεύω να έχω φαντάζομαι ότι θα έχω προβλήματα με ορισμένε από τι τροπολογίε μου και χωρί να έχω μυρίσει τα δάχτυλά μου είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνεί με τη 36-161. Θα έλεγα υπάρχει μια συνοχή όμω μεταξύ των τεσσάρων τροπολογιών. Και όχι επειδή η Περβάος Περέζα ε, ενδιαφέρεται για τους ε, οίκους αξιολόγησης ότι θα πρέπει να φανταστούμε σημεία και τέρατα. Παγκοσμίως, στην εποχή των ε, πιο εξεζητημένων τεχνολογιών ε, της πληροφορικής κλπ. Όταν στέλνετε μία συστημένη επιστολή στις Βερμούδες ή όταν ε, μέσω ίντερνετ παραγγέλνετε ένα μπουλόνι το οποίο έχει φτιαχτεί στην Ταϊβάν, μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο όλη την διαδικασία αυτών, κίνησης αυτών των προϊόντων. Πότε έχει εκδοθεί το τιμολόγιο, πότε τυλίχτηκε, πότε συσκευάστηκε, πότε το φόρτωσαν στο βαπόρι. Αλλά και εδώ και στο δικό μας τον τομέα μπορεί να είναι χρήσιμη η σύγχρονη τεχνολογία. Στις Ηνωμένε Πολιτείες και στα πλαίσια του πακέτου Dodd-Frank συζητιέται για το πώς μπορούμε να έχουμε ανιχνευσιμότητα στην διακίνηση κεφαλαίων. Αυτό ενδιαφέρει τους, ε, τα στελέχη των επιχειρήσεων όταν θέλουν ε, να διαπραγματευτούν μια επιχειρησιακή στρατηγική και δεν γνωρίζουν ε, τα κεφάλαια των συμμετεχόντων. Οι Αμερικάνοι θέλουν λοιπόν να προχωρήσουν σε αυτή την ανιχνευσιμότητα των κεφαλαίων που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να προσέξουμε να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση που είχαμε βρεθεί τότε με τη λογιστική καταγραφή κάποιος ξεκινάει μια διαδικασία σε εθνικό επίπεδο στην άλλη άκρη του πλανήτη ε, ενώ το θέμα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια παγκόσμια ανιχνεσιμότητα όπως χρειαζόμαστε και ένα παγκόσμιο λογιστικό σύστημα και αν η Ευρώπη δεν ανέβει στο τρένο αυτό γρήγορα, τότε οι Αμερικάνοι θα προχωρήσουν από τη μεριά τους και κάποια μέρα θα έρθουν εδώ και θα πούνε ορίστε αυτή είναι η ανιχνευσιμότητα των κεφαλαίων, έτσι γίνεται, έχουμε ορίσει ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι κανόνες, Λοιπόν, ή παίρνετε ή αφήνετε τελείωσε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν άλλους τρόπους. Γι' αυτό πρότεινα την τροπολογία 161 με τις ευλογίες ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ελπίζω να με υπερασπιστείτε, να τη δεχτείτε. Τώρα τα δύο πακέτα έχουν σχέση με την 30 με την 3777 Αυτοί που έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένε εργασίες στον τομέα και ιδιωτικοποίησαν αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι του δημοσίου τομέα είναι η οίκη αξιολόγησης. Θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε την διατύπωση, πρέπει όμως να αναφερθεί και η μία συμπληρώνει την άλλη. Και με αυτά που είπε ο κύριος ε, Τρέμοσάη. Να θυμάστε τι έχει εγκρίνει και το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της Επιτροπής ε, Κρίσης, ούτως ώστε να μην αντιφάσκουμε. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να έχουμε μία ολοκληρωμένη παγκόσμια διακυβέρνηση μέσα από τις ε, γραμμές ε, του G20 γνωρίζουμε όλοι τους μηχανισμούς, ο συνάδελφος αναφέρεται σε αυτό, αλλά για να ξεπεράσουμε όμως αυτό το κάπως ε, βρεφικό στάδιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης πρέπει να προσετεριστούμε το G20 όπως και τις διαρθρώσεις της οικονομικής διακυβέρνησης που εξεργαστήκαμε σε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και του ΟΗΕ. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Κρίσης ε, για αυτό το σημείο μας βοηθούν να προχωρήσουμε. Το δεύτερο σημείο, συμπληρωματικό σημείο, είναι η διακίνηση των κεφαλαίων. Στην έκθεση της Επιτροπής ε, Κρίσης λέμε ότι η Επιτροπή Εποπτείας δεν θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο περιμένοντας την επάνωδο στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και την λειτουργία τους έναντι των μακροοικονομικών στόχων. Αν δηλαδή η διακίνηση των κεφαλαίων επιβαρύνει την ε, ε, αστάθεια την αστάθεια, τότε ε, ο ρόλος εμπίπτει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα, συγγνώμη, δεν θυμάμαι εγώ ακριβώς όλες τις τροπολογίες, αλλά είναι δύσκολο να μιλήσουμε για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση χωρίς να αναφερθούμε στους οργανισμούς αυτορύθμισης ή στους, ε, στον ιδιωτικό τομέα. Επιτροπή της Βασιλείας ή την ESB. Τώρα για την Επιτροπή της Βασιλείας έχουμε πολλές ε, τροπολογίες. Αλλά στο τελικό κείμενο του ψηφίσματος θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να αναφερθούν διότι ανήκουν στο πακέτο της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ Περβόνς. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης ηγετής. Αλλά ο Σαΐτ Καμάλ μου ζήτησε να τον αναπληρώσω, γιατί ψηφίζει αυτή τη στιγμή σε άλλη επιτροπή. Πάντως, πολύ ευχαρίστως να τον αντικαταστήσω και να διαβάσω τα σχόλιά του. Θερμές ευχαριστίες καταρχήν εκ μέρους του κόμματος των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερος που μια τόσο ευαίσθητη έκθεση βρίσκεται σε λογικά χέρια και την έχει αναλάβει ο αξιότιμος Γκένορ Χέκμαρκ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που συνεργαζόμαστε μαζί του. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι δυνάμεθα και θα οφείλαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο, ε, παγκόσμιο όργανο επίσημο μέσω στη δομή και χέγγε και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του Γκέναρ ε, προσοχή όμως ε, να μην δώσουμε στον κίνδυνο της ε, υπερβολικής ρύθμισης. Πάντως έχω διαπιστώσει ότι έχουμε παρεμφερήσεις απόψεις με τον Γκέναρ Χέκμαρκ για το θέμα αυτό. Να αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Πολύ σημαντική λοιπόν η θέση τους. Θα πρέπει να λάβουμε αυτή τη σημασία υπόψη και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα, και το τονίζω αυτό, όλα τα υπάρχοντα μέσα συνεργασίας, όπως το, διάλογο, το διατλαντικό διάλογο νομοθετών και άλλες μορφές συνεργασίας, να χρησιμοποιήσουμε τα χιστάμενα μέσα και να ενθαρρύνουμε και οι διεθνείς οργανισμούς όπως το G20, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, να μειώσουν τα ελλείμματα, να έχουν καλύτερη συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα που αντιλήσαμε τους τελευταίους μήνες και χρόνια. και κατά τη γνώμη μου δεν θα σας εκπλήξει ότι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και σκεπτικιστές ό,τι αφορά το φόρο ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Και είμαστε επιφυλακτικοί κατά οποιοδήποτε επιπρόσθετου φόρου. Δεν θα υποστηρίξουμε τίποτα σχετικό. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα σχόλια ως προς την έκθεση του Γκίνορ και τον ευχαριστώ θερμά για την μεγάλη του προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε, Κλούτε. Να ευχαριστώ. Και εγώ δεν είμαι σκιώδης. Ο Μιγγέλ Πόρτας είναι από την ομάδα μας, αλλά έχει αλλού υποχρέωση μου έγραψε κάποιες σημειώσεις και μου ζήτησε να τις διαβάσω. Και αυτό θα κάνω, τα έχει κάνει στα αγγλικά, οπότε και εγώ θα τα διαβάσω στα αγγλικά. Και μετά θα κάνω και τις δικές μου παρατηρήσεις. Ξεκινήσω με αυτά τα οποία μου έχει δώσει ο Μιγγέλ. Ο Γκούναρ θεωρεί πως οι ανισορροπίες εμφανίζονται λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας των οικονομιών. Εμείς θεωρούμε πως η ανταγωνιστικότητα δεν θα πρέπει να είναι το βασικό ζήτημα της οικονομίας. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας δεν είναι η αιτία αλλά η συνέπεια της παγκόσμιας οικονομίας που υφίσταται τον νόμο του ισχυρού χωρίς ε, συνεργασία. Πρώτα απ' όλα στο εκτιμώντας και στην παράγραφο 13 επιμένει ο Γκούναρ στην σημασία του ελευθέρου εμπορίου για την ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε πως το ελεύθερο εμπόριο είναι προστατευτισμός υπέρ των πλουσίων. Οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες εξάγουν προϊόντα ε, εκεί που έχουν περισσότερα πλέον εκτήματα. Χρειάζεται μια άλλη στρατηγική με βάση το δίκαιο εμπόριο. Το δίκαιο εμπόριο στηρίζει εκείνους που πρέπει να υποστηριχθούν. Δεν είναι προστατευτισμός, προσπαθεί να επιτύχει έναν συντονισμό ε, καθώς ε, ελλείμματα και πλεονάσματα είναι πτυχές του ίδιου προβλήματος και βεβαίω καταπολεμά τον ανταγωνισμό που βασίζεται στου χαμηλού μισθού και τη φοροδιαφυγή. Δεύτερον, η δεύτερη διαφωνία είναι θεσμική. Ο Γκούναρ θα ήθελε στο Δουνουτού να πάει η παγκόσμια διακυβέρνηση. Εμείς ε, ασκούμε κριτική στην έλλειψη δημοκρατίας του G20, G7 και G8, αλλά το να ε, δοθούν σε αυτού του τραπεζίτε οι δυνατότητε διακυβέρνησης ταυτόχρονα δημιουργεί προβλήματα στις ε, χώρες και είναι αντίθετο με κάθε έννοια της δημοκρατίας και της ισότητας μεταξύ των κρατών. Ο συντονισμός θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της, ε, των δομών του ΟΗΕ και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του. Πρέπει να δούμε μια περιφερειοποίηση της παγκοσμιοποίησης με περιφερειακές συμφωνίες θα βασίζονται σε μακροοικονομικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δίκτους. Αυτά ήταν τα σχόλια του Μιγγέλ Πόρτας. Εγώ ίδιος θα ήθελα να προσθέσω, να υπενθυμίσω πως είναι για μένα έχει μεγάλη σημασία τροπολογία 69 που έχω καταθέσει και αφορά το ζήτημα της κερδοσκοπίας με πρώτες ύλες και τρόφιμα και θα ήθελα εδώ πέρα να έχουμε έναν συμβιβασμό που θα τον δεχτεί η πλειοψηφία. Νομίζω πως είναι ένα θέμα που τουλάχιστον στον τύπο που διαβάζω εγώ παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Στο είδαμε και το θίξαμε στις τελευταίες συζητήσεις με τον Μισελ Μπαρνιέ και είναι καιρό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να καταλήξουμε σε ένα λογικό συνδυασμό εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με πολλές από τις ε, συστάσεις ε, του εισηγητή. Νομίζω πως και κάποιες τροπολογίες μπορούν να ξεκαθαρίσουν τα βασικά μηνύματα της έκθεσης. Τώρα έγινε μια διάκριση μεταξύ ουσίας και θεσμικών ζητημάτων. Επί της ουσίας μπορούμε να πούμε πως η Κομισιόν συμμετέχει στις συζητήσεις για την παγκόσμια διακυβέρνηση στα κατάλληλα φόρα, στην ομάδα των 20 που κυρίως αναφέρθηκε, τονίζουμε την ανάγκη καλύτερου παγκόσμιου μακροοικονομικού συντονισμού, κυρίως στο πλαίσιο των G20 για ισχυρή πολυμερή ανάπτυξη, για να δούμε παγκόσμιες διαχείρισης αποτελεσμάτων θεωρούν πως το τωρινό νομισματικό σύστημα δεν έχει ένα μηχανισμό εξορρόψης ε, και ειδικά έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής. Οπότε η ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας και στο επίπεδο του Δονοτού και στους G20 έχει κέρια σημασία. Όσον αφορά τη διαχείριση των παγκοσμίων ροών κεφαλαίου που επίσης ζήτησαν οι G20 θεωρούμε πως πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και θα πρέπει να αναπτύξουμε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές όμως θα πρέπει αυτό να αποτελέσει τελευταία λύση Θεωρούμε πως ε, τα πρωτογενή αυτά μέσα θα πρέπει να παραμένουν οι σωστές ε, κατάλληλες δομές. Τώρα για τα ειδικά τραπεζικά δικαιώματα και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στο διεθνές σύστημα. Πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα τον κίνδυνο ενός πολυπολικού συστήματος Οι παρατηρήσει αυτές κατέθηκαν και στους G20. Και η κυρία Μπέρες επίσης ανέφερε το θέμα των σχέσεων μεταξύ των G20 και του ΟΗΕ. Και, όπως ξέρετε, ξεκίνησε μια συζήτηση στον ΟΗΕ μετά την ε, εντολή του 65-94 του ψηφίσματος Γενικής Συνέλευσης για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και η οικονομική, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα. Επίσης υπάρχει στο Σαντιάγο της Χιλής ε, ε, σεμινάριο σήμερα ακριβώς για αυτό το θέμα. Για τα θεσμικά τώρα να ολοκληρώσω με κάποιες παρατηρήσεις για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στην ε, συζήτηση περί οικονομικής πολιτικής. Θεωρούμε πως ε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή φόρα είναι κρίσιμος παράγοντας, ειδικά για να μιλήσει με μία φωνή. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκπροσωπείται ε, ως τέτοια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι απλώς παρατηρητής, ενώ σε άλλα διεθνή φόρα που επίσης αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης, η κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι ιδεώδης. Επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Μετά την θέση ενισχύ ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι μεταβατικές διατάξεις φαίνεται πως δεν βελτιώνουν την εκπροσώπηση και το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουν στο status quo. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, ειδικά όπως ε, ανέφερε ο Επίτροπος ο κύριος Ρέν στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 6 ε, Ιουνίου. Είπαμε πώς είναι προς το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να πάνε σταδιακά σε μία ε, θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα για την προσέγγιση που θα θέλαμε θεωρούμε ε, καθαρά σε νομοθετικούς όρους πως η επέκταση της νομοθεσίας ε, στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και επιτήρησης όπως προγραμματίζεται από το Συμβούλιο θα πρέπει νομίζουμε να οδηγήσει σε μια ενιαία εκπροσώπηση της Ένωσης σε διεθνείς τέτοιους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 17 της Συνθήκης περί άσκησης εσωτερικών αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα είναι εύκολο να προτείνουμε μία ενιαία εκπροσώπηση σύμφωνα με το άρθρο 17 ως προείπα. Όπως βλέπετε λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η συζήτηση όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχει για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και πάλι επιβεβαιώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή, σχεδόν και την Επιτροπή και ιδιαίτερα καλωσορίζουμε την ακρόαση που θα γίνει με το ίδιο θέμα στις 27 Ιουνίου και αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, ευχαρίστω να δώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τις απόψεις που παρουσίασαν. Έχω δύο γενικέ παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου που συζητούμε τι θέλουμε να μην περιληφθεί στη διαδικασία αυτή και πού θα θέλαμε να οδηγεί αυτή η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Γιατί μερικές φορές όταν μιλούμε για παγκόσμια διακυβέρνηση έχω την αίσθηση ότι κάποιοι συνάδελφοι υπενήσονται ένα είδος παγκόσμιας οικονομικής κυβέρνησης. Αυτό αποκλείεται, είναι ανέφικτο. Έτσι όμως θα, έχουμε την ευκαιρία, θα, θα χάσουμε την ευκαιρία να ασκήσουμε και την επιρροή σε ορισμένα θέματα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Παρακαλώ να επικεντρωθούμε στο εφικτό, στο δυνατό σε παγκόσμιο επίπεδο και να μην ξεφεύγουμε σε πράγματα τελείως ανέφικτα. Μερικές φορές θα μιλούμε για την παγκόσμια οικονομία. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν τις τελευταίες δεκαετίες ως ε, ολέθριες. Δεν συμφωνώ. Δεν ισχύει αυτό. Οι τελευταίες δεκαετίες ήταν ε, μεταβολή προς το καλύτερο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι αναφέρθηκε αυτό. Το πρόβλημα έγκυται στη ραγδαία μεταβολή της δομής παγκόσμιας οικονομίας. Γιατί σχετικά πρόσφατα η παγκόσμια οικονομία ήταν ουσιαστικά οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Δυτική Ευρώπη. Και πολλά, πολλές παγκόσμιες οργανώσεις σε αυτή τη διάκριση στηρίζονται. Το είπαμε και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να τη διοικούν οι Αμερικανοί και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο οι Ευρωπαίοι. Αυτά στο πρόσφατο, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, αλλά τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει. Η κατάσταση έχει μεταβληθεί ριζικά και έχουμε νέε προκλήσει. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ο κύριο Εκλιούνα είπε ότι έχουμε δει μια μεγάλη χρηματοπιστωτική διαφορά τα τελευταία χρόνια και μια κατάρρευση. Το θέμα είναι πώ θα αναχαιτήσουμε ή θα αποτρέψουμε αντίστοιχη κατάρρευση και στο μέλλον. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε. και όταν μιλούμε για τα διάφορα σκέλη της έκθεσης. Ένας λόγος των πλεονασμάτων στην παγκόσμια οικονομία είναι τα ελλείμματα επίσης στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί δεν υπάρχει πλεόνασμα χωρίς έλλειμμα. Και πολύ συχνά τα ελλείμματα ε, οφείλονται στις εθνικές πολιτικές. Όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά, αν κοιτάξουμε την αμερικανική οικονομία για παράδειγμα. Βέβαια, οι δεκαετίες χαλαρής σχετικά νομισματικής πολιτικής επηρέασε τα πράγματα και συνέβαλε στο έλλειμμα της ε, ε, αμερικανικής οικονομίας σε αντίθεση με το πλεόνασμα της κινέζικης οικονομίας. Είναι αλληλέδετα τα ελλείμματα με τα πλεονάσματα. Οπότε αυτή την άποψη είναι σημαντικό στην παγκόσμια δικυβέρνηση να έχουμε νομισματικές πολιτικές και να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτές επηρεάζουν το γενικό πλαίσιο. Και φυσικά η, τα ελλείμματα στα, δημόσια οικονομικά φυσικά επηρεάζουν και την υπόλοιπη κατάσταση. Το βλέπουμε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι κεντρικά ζητήματα και σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο. Επίσης ε, μιλάμε για τις ε, για τους διάφορους οργανισμούς, τα διάφορα θεσμικά όργανα. Όλα αυτά τα όργανα, είτε είναι τυπικά είτε άτυπα, έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αναφέρθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο επίπεδο για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Εκτός αν είχαμε κάτι αντίστοιχο <laughs> με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ για τα οικονομικά, νομίζω δεν θα, θα ήταν καταστροφικό κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συμφωνώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες δομές. Και το G20 είναι σημαντικό. Λόγω του μεγέθου των οικονομιών των χωρών που συμμετέχουν εκεί. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και αυτή η επιλογή είναι πολύ αυθαίρετη. Η Σουηδία και η Μάλτα δεν συμμετέχουν στου G20 αλλά δεν μόνο εκεί το πρόβλημα. Είναι αυθαίρετη η επιλογή, γιατί και άλλε οικονομίε θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στους 20. Και μερικέ από αυτές που συμμετέχουν στου 20 θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι εκτό. Επίση θα πρέπει να δούμε για... με τι κριτήρια προσδιορίζουμε την ισχύ μια οικονομία. Χαρακτηρίζουμε μερικέ οικονομίε ω μεγάλε. Τι γίνεται με τι αναδυόμενε οικονομίε, Μήπω θα πρέπει να τι λάβουμε καλύτερα υπόψη. Επίσης, ε, μήπως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ε, οικονομίες που τη χάνουν διαχείριση σχέση με άλλες που έχουν χειρότερη διαχείριση. Αυτά για ορισμένα προβλήματα που μερικές φορές αποφεύγουμε να συζητήσουμε. Το G20 πάντως εξορισμού είναι σημαντικό όργανο και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχει όμως πρόβλημα εφαρμογής στο G20 σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς παραδείσους που αναφέρθηκαν. Οι κεφαλαϊκές απαιτήσει ή διάφορα άλλα κριτήρια. Να βρούμε ένα είδος συνύπαρξης μεταξύ G20, Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου και άλλων οργάνων τυπικών και ατύπων θα ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω. Και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία αν θέλουμε να ρυθμίσουμε την οικονομία, αλλά στόχος μας, στόχος μας είναι να θέσουμε κάποια πλαίσια στην παγκόσμια οικονομία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, άλλο το πλαίσιο και άλλο η ρύθμιση. Και αυτό το διαχωρισμό θα πρέπει να τον εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ ε, και την Προεδρία που επέτρεψε τη διεξαγωγή αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή. Επιτέλους, καλό αργά παραποτέ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ξαναλέω ότι τη Δευτέρα 27 στις 4 το απόγευμα θα έχουμε μία ακρόαση για το θέμα με τους προσκεκλημένους που ήδη γνωρίζετε. Θα ψηφίσουμε σε αυτήν την Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσουμε μετά στην Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κλείνω με αυτό το σημείο. Διάφορα, όχι. Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 27 Ιουνίου. Ολοκληρώσαμε.